Περνάμε στο δέκατο της ημερήσιας διάταξής μας σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στη διάσκεψη του Βερολίνου. Εφαρμογή του εμπάργου όπλων στη Λιβύη. Στο θέμα αυτό έχουμε προσκαλέσει και μέλη της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέπ και καλωσορίζω τα μέλη αυτά στη σημερινή συνεδρίαση. Επίσης θα ήθελα να καλωσορίσω τις δύο ομιλήτριές μας, την κυρία Στεφανή Βίλιαμς από τα Ηνωμένα Έθνη, η οποία λόγω της συνεδρίασης των 5 συν 5 της Κοινή Στρατιωτικής Επιτροπής για την Εκεχηρία στη Λιβύη βρίσκεται στη Γενέβη και θα συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης μαζί μας. Και βεβαίως να καλωσορίσω και τη Ρόζα Μαρία Τζιλ, επικεφαλής της ομάδας για τις χώρες του Μαγκρέπ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράση. Στη συνέντευξη του ο στρατηγός Γκρατσιάνο, πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ένωσης, αναφερόμενος στη Λιβύη, σημείωσε πως στη μακρά του καριέρα δεν έχει ξαναδεί έναν πραγματικό πόλεμο τόσο κοντά στα σύνορα της Ένωσης. Λίγο πριν, στη συνεδρία στη ΣΕΝΤΕ, συζητούσαμε για την κατάσταση ασφάλειας στο Μάλι, όπου μία από τις αιτίε για την κρίση εκεί είναι το λαθρεμπόριο όπλων από τη Λιβύη. Η απόφαση για το εμπάργκο όπλων έχει αποφασιστεί με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ήδη από το 2011. Η ανάγκη εφαρμογής της συγκεκριμένη απόφασης από όλους τους εμπλεκόμενους επιβεβαιώθηκε και στην πρόσφατη σύνοδο του Βερολίνου. Όμως, όπως δήλωσε και χθε ο ύπατος εκπρόσωπος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μπορέλ, αυτό δεν έχει συμβεί η επιχείρηση Σοφία, όπως αργότερα ονομάστηκε από το όνομα ενός κοριτσιού που γεννήθηκε στη γερμανική φρεγάτα, ξεκίνησε το 2015 με κύριο στόχο την καταπολέμηση των κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων και από το 2016 συμπεριλήφθη η εκπαίδευση της Λιβικής Ακτοφυλακής και τήρηση του εμπάργου όπλων. Όμως τον τελευταίο καιρό η ναυτική αυτή επιχείρηση δεν έχει πλοία. Χθε, στη συνεδρία του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών, αποφασίστηκε η ανάληψη νέα στρατιωτική επιχείρηση στα νυχτά τη Λιβύη, η οποία θα αντικαταστήσει την επιχείρηση Σοφία και στόχο θα έχει την εφαρμογή του εμπάργου όπλων που έχει αποφασίσει το Συμβούλιο Ασφαλεία του ΟΗΕ. Οι λεπτομέρειε, όπω φαίνεται, θα αποφασιστούν στην επόμενη συνεδρία των Υπουργών Εξωτερικών. Έχοντα υπόψη όλα αυτά, θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα στην κυρία Βίλιαμ για 10 λεπτά για να μας ενημερώσει που βρισκόμαστε σχεδόν ένα μήνα μετά τη Σύνοδο του Βερολίνου. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα. Χαίρομαι που ήρθα να μιλήσω από τη Γενέβη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου μόλις σήμερα ξεκινήσαμε το δεύτερο γύρο των ε, νέων ομιλιών 5 5 μεταξύ των διαφορών μερών ε, της ε, διένεξης της στη Λιβύη, της διαμάχης στη Λιβύη και σήμερα συνεχίζονται αυτές οι ομιλίες ε, μαζί με την ανακτήρια συναντήση της Διεθνούς Επιτροπής για την Λιβύα, Λιβύη μετά από τη διασκέψη του Βερολίνου. Η πρώτη συνάντηση AFCO έλαβε χώρα στο Μόναχο μόλις πριν δύο μέρες. πιστεύω είχε θετική έκβαση. Έγιναν σοβαρές ε, συνομιλίες. Ε, βάσει των ε, συμπερασμάτων της διάσκεψης του Βερολίνου και των προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, καθώς υλοποιούμε όχι μόνο τα συμπεράσματα του ανακοινωθέντος του Βερολίνου, που συνολικά πιστεύουμε αντιμετωπίζει τα προβλήματα που υπάρχουν στη Λιβύη και που είναι περίπλοκα, αλλά και το ψήφισμα που υιοθετήθηκε στα Ηνωμένα την περασμένη εβδομάδα, το ψήφισμα 25-10 που υποστηρίζει τα συμπεράσματα της διάσκεψης του Βερολίνου. Τι πέτυχε η διάσκεψη του Βερολίνου ε, πολύ θετικά τη δημιουργία ε, ενός διεθνούς μηχανισμού προστασίας ε, ε, για τη Λιβύη στο πλαίσιο του οποίου θα λειτουργεί η Ανσμιλ. Από τον Ιανουάριο του 19 μέχρι σήμερα, αν δει κανείς τι έχουμε κάνει εμείς ε, για να υλοποιήσουμε το επιχειρησιακό έγγραφο που συνόδευε τη διάσκεψη του Βερολίνου, η Ανσμιλ ε, συνέθεσε και παρουσίασε στις 13 ε, χώρες και στις ε, τρεις περιφερειακές οργάνωσεις που συμμετείχαν στο Βερολίνο το δικό μας όραμα για το πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τα συμπεράσματα της διάσκεψης, να τα υλοποιήσουμε. Να περάσουμε δηλαδή από μια διεθνή διαδικασία σε μια λιβική διαδικασία. που σχετίζεται με την πρόταση του ειδικό απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα, του κ. Σαλάμα. Ε, έγιναν πολλές σημαντικές συναντήσεις, η μία στην Αλγερία, όπου η Αλγερία κάλεσε μια υπουργική με τους γείτονες τον Ιανουάριο του 2013 μετά η Αφρικανική Ένωση ε, διοργάνωσε μια επιτροπή ψηλού επίπεδου στις 30 Ιανουαρίου ε, στην ε, Δημοκρατία του Κονγκό και μετά έγιναν συνομιλίες στην 33η Τακτική Σύνοδο τη Σύνοδου Κορφής ε, της Αφρικανικής Ένωσης ε, ε, τον Φεβρουάριο και μετά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης χθες εδώ στις Βρυξέλλες. Υπάρχει λοιπόν η τακτικη συνοδο τη συνοδου της αφρικανικης ενωσης τον φεβρουαριο και μετα το συμβουλιο αυτή και διεθνής προσοχή συνδέεται με το ψήφισμα 2510 10 μήνες μετά από σχετική αδράνεια από το Συμβουλίο Ασφαλείας. Εκεί υποστήριζεται σαφώς η έκκληση για ε, διαρκή χειρία. Το ψήφισμα είναι σημαντικό γιατί χρειαζόταν οι Λίβοι να ακούσουν κάτι τέτοιο από το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι υπάρχει αυτό το μήνυμα. Ότι η χώρα έχει, βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής της διεθνούς κοινότητας και ότι υπάρχει υποστήριξη για την ειρηνική τη σταθερότητα, κάτι που επιθυμούν πολύ λίγοι φυσικά. Τι έχουμε κάνει εμείς και πριν τη διασκέψη του Βερολίνου και μετά από αυτήν. Δραστηριοποιήσαμε και τις ε, τρεις λύσεις ε, του εγγράφου μας ε, οικονομική, ασφαλείας και πολιτική. Την οικονομική λύση την είχαμε ενεργοποιήσει πριν το Βερολίνο στις 6 Ιανουαρίου. Είχαμε συγκαλέσει οι εμπειρογνώμονες για να ξεκινήσουν συζητήσεις για τη δημιουργία δύο επιτροπών. Η μία αφορά εμπειρογνώμονες σε οικονομικά θέματα για τη Λιβύη και η άλλη ένας μηχανισμός για την ανάπτυξη και την ανοικοδόμηση. Η Επιτροπή Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων Μόλις την περασμένη εβδομάδα στο Κάιρο συνεδρίασε για δεύτερη φορά μετά από δική μα σύγκληση και αυτοί ενέκριναν και συμφώνησαν το σχέδιο ε, του τρόπου εργασία αυτή τη Επιτροπή ε, και ε, περιγράφεται εκεί ποια θα είναι τα κατεπήγοντα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί η Επιτροπή, εστιαζόμενη στα άμεσα προβλήματα τη Λιβύη όσον αφορά την οικονομία και το τραπεζικό σύστημα, που αυτή τη στιγμή δέχονται τεράστια πίεση λόγω του προβλημάτων με το πετρέλαιο και της ανωτέρας βίας, ουσιαστικά το κλείσιμο της ε, παραγωγής πετρελαίου στη Λιβύη, που ήταν η μόνη πηγή ε, εσόδων για το Λιβικό κράτος. Επίκυνται λοιπόν πιθανώς ε, ε, σημαντικά προβλήματα και μια σοβαρή ενδεχομένω τραπεζική κρίση λόγω φερεγγιότητα πολλών τραπεζών στη Λιβύη μέσα στους επόμενους μήνες ε, συμπεριλαμβανομένη της μεγαλύτερης τράπεζας ε, στη χώρα κάτι που θα οδηγήσει σε κοινωνικά, οικονομικά προβλήματα στον πληθυσμό. Έχουμε σχηματίσει τρεις ε, ομάδες εργασία μετά από αυτή την δεύτερη συνεδρία στο Κάιρο. Μία η οποία θα ασχοληθεί με κάποια από αυτά τα ζητήματα ε, όσον αφορά τη διακοπή της ε, πετρελαιοπαραγωγή, την κατανομή των εσόδων, την αποκέντρωση, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη διαφάνεια. Αυτό είναι ένα σύνολο προβλημάτων. Ένα δεύτερο σύνολο προβλημάτων είναι η κρίση του τραπεζικού τομέα που βρίσκεται ουσιαστικά στο επίκεντρο των θεσμικών ε, διχασμών ε, στη χώρα, το διαχωρισμό της κεντρικής τράπεζας Λιβύας σε ένα ε, τμήμα στην Τρίπολη και σε ένα άλλο τμήμα στην Ανατολική Λιβύη. Η τελευταία ομάδα εργασία θα εστιαστεί στην ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη. Ανοικοδόμηση, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι αφού θα διασφαλιστεί ε, ειρήνη και σταθερότητα, τα έργα ανοικοδόμησης θα κατανεμηθούν ισότιμα στη χώρα, διότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς πολλές πόλεις έχουν καταστραφεί σημαντικά στην Ανατολική Λιβύη και στο Νότο και φυσικά τώρα πλέον και στη Δυτική Λιβύη, την ευρύτερη περιοχή της Τρίπολης, την Βοσεφάνα που έχουν επίσης καταστραφεί ε, αυτή η τελευταία καταστράφηκε το 2014. Και φυσικά είχαμε και τις πρώτες στρατιωτικές ομιλίες εδώ στη Γενέβη που έλαβαν χώρα μεταξύ 3 ε, ε, και 8 Φεβρουαρίου. Μια εξαήμερη συνάντηση που αποτέλεσε ένα πρώτο βήμα για να διασφαλιστεί μια διαρκή εκεχηρία ενισχύει και βασίστε στην ε, ε, πάυση του πυρός που είχε επιτευχθεί με την πρώτη συνάντηση. Ήταν πολύ επικοδομητικός ο πρώτος γύρος. Οι δύο αντιπροσωπείες αποφάσισαν να μην συναντηθούν ε, άμεσα. Διεξήγαμε λοιπόν παράλληλες διαπραγματεύσεις και επιτύχαμε τη διατήρηση της εύθραυστης εκεχηρίας που απαιτείται επίγοντος για να διασφαλιστεί η εδαφική ακαιρεότητα της Λιβύης ε, και για να φύγουν οι μη Λιβύοι μαχητές και για να διασφαλιστεί η καταπολέμηση των τρομοκρατικών ομάδων. Επίσης, συμφώνησαν και οι δύο πλευρές ε, για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως η ε, ανταλλαγή κρατουμένων και σωρών Αναφέρθηκε η ανάγκη επιστροφής στα σπίτια του των εκτοπισμένων, αλλά αυτό φυσικά αφορά ζητήματα εκεχηρία. Μπορεί κανείς να διαχωρίσει δυνάμεις ε, ή ενδεχομένω να υπάρχει μια ειρηνική περιοχή όπου, μέσω τη οποία μπορούν οι άνθρωποι να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Γι' αυτό ξαναξεκινήσαμε σήμερα τις διαπραγματεύσεις, ούτως ώστε να επιτύχουμε κάποια εκεχηρία έχουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορες δυσκολίες επιτόπου. Έχουμε πάνω από 200 ε, παραβιάσεις της ε, εκεχήρίας της 12 ε, Ιανουαρίου. Παρακολουθούμε φυσικά την εκεχηρία. Ο μηχανισμός παρακολούθησης θα πρέπει να αποφασιστεί στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας σε αυτή την κοινή στρατική επιτροπή στη διαδικασία 5 5, αλλά είχαμε διάφορες παραβιάσεις της Παυστουπυρός και σήμερα μάλιστα ε, όπου ε, είχαμε το ε, στο, επίθεση με πυράβλους στο λιμάνι της Τρίπολης και μάλιστα σε ένα δεξαμενόπλιο που ξεφόρτωνε υγροποιημένο φυσικό αέριο. αν αυτό το πλήσιο είχε πληγεί, τότε η τραγωδία θα ήταν τεράστια. Ε, χρησιμοποιούνται λοιπόν ε, ε, τεθωρακισμένα και πύραυλοι. Έχει πληγεί το λιμάνι, το αεροδρόμιο. Υπάρχουν συγκρούσεις σε διάφορες περιοχές στα ανατολικά της Τρίπολης, στην Βουενγκρέιν και στην Βόσκα. Παραμένουν λοιπόν έντονες εντάσεις στην πρώτη γραμμή. Δεδομένων αυτών, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να υπόσχονται ότι θα κάνουν μια προσπάθεια να διατηρήσουν την εκεχηρία. Το άλλο φυσικά που παρατηρούμε με μεγάλη ανησυχία και πιστεύω το έχουμε πει πολύ καθαρά δημοσίως ότι είναι απαράδεκτες οι καταφορές παραβιάσεις του εμπάργου όπλων των ΗΕ. Γι' αυτό καλωσορίζουμε την απόφαση που ελήφθη χθε ε, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι αναγκαίο ως πρώτο βήμα, διότι η Λιβύη ουσιαστικά είναι γεμάτη όπλα, δεν χρειάζεται άλλα όπλα. Εσείς κύριε Πρόεδρε αναφερθήκατε σε όπλα τα οποία φεύγουν τώρα πια, περνάνε από τα σύνορα της Λιβύης όπως περνούσαν εδώ και χρόνια και ε, θέτουν σε κίνδυνο και τις χώρες του Σαχέλ, ε, τις εκθέτουν σε αυξημένη τρομοκρατία και βία. Φυσικά η ανθρωπιστική κατάσταση ε, την παρακολουθούμε πολύ στενά διότι οι απλοί άνθρωποι στη Λιβύη βλέπουν τη ζωή τους να επιδεινώνεται ένα στους τέσσερις ε, ε, και παραπάνω έχουν πλέον επηρεαστεί αρνητικά από τις διαμάχες. Η μισή από το 1,8 εκατομμύρια ανθρώπους ε, που έχουν πληγεί από την κρίση στη Λιβύη χρειάζονται κάποιο είδου ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό σημαίνει σχεδόν το 1 τρίτο των μη Λίβιων μεταναστών και προσφύγων. Αυτέ οι επιθέσει σε άμαχου πληθυσμού και σε υποδομέ ε, μη στρατιωτικέ, ε, ειδικότερα και στην Τρίπολη, έχουν διπλασιαστεί τέτοιε επιθέσει το 2019 μετά από την επίθεση στην Τρίπολη στις 4 Απριλίου που είχε ως αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς πάνω από 149.000 άνθρωποι ε, αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια του στην περιοχή της Τρίπολης μετά από τότε που ξεκίνησε τον Απρίλιο η διαμάχη και σχεδόν 345.000 άνθρωποι παρέμειναν, έμεναν σε ε, περιοχές της πρώτης γραμμής και εξακολουθούν να διατρέχουν ε, κίνδυνο εκτοπισμού. Συγγνώμη πρέπει να... Ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Λοιπόν, θα κλείσω λέγοντα ότι έχουμε δεσμευτεί να συνεχίσουμε ε, στις τρεις αυτές οδούς. Έχουμε ανακοινώσει την έναρξη του πολιτικού διαλόγου που επίσης θα λάβει χώρα στη Γενέβη ξεκινώντας στις 26 Φεβρουαρίου. Στο Λιβικό Κοινοβούλιο υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες και εμείς απευθύνουμε έκκληση ουσιαστικά στο Κοινοβούλιο να δράσει και να τηρήσει μια διαφανή δημοκρατική διαδικασία ε, για να εκλέξει, για να επιλέξει τους εκπροσώπους της ε, συναντήσεις αυτές. Εμείς έχουμε τη δική μας ποσόστοση για αυτή τη συνάντηση και θα χρησιμοποιήσουμε τη δική μας ε, ποσόστοση φυσικά, ούτως ώστε να ίσως ισοτιμία ε, ίση εκπροσώπηση φιλών, μειονοτήτων και οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών. Σε αυτή τη συνάντηση εδώ στη Γενέβη, σε 9 μέρες από τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα σταματήσω εδώ.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 We consider that the EU is a is expected to play a role in Libya, a much stronger role than what we, we have been able to play so far. And we think that there is now... Και υπάρχει αυτή η κατάσταση τώρα για δύο λόγους. Τον ένα το έθιξε η Στεφανή. Είναι μια νέα διαδικασία αυτό που συνέβη στο Βερολίνο και η συνέχεια που δόθηκε, η συνέχεια μετά το Βερολίνο. Το δεύτερο είναι το μήνυμα ενότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λιβύη, για το θέμα της Λιβύης. Για το Βερολίνο. Πιστεύουμε ότι το Βερολίνο έκανε κάτι πολύ σημαντικό. Σε μια πολύ σημαντική χρονική στιγμή. Σε μια στιγμή όπου η Λιβύη έβλεπε ότι υπήρχε πολλαπλασιασμός επικίνδυνων πρωτοβουλειών. Ο ΙΕ είχε την ιδέα, μετά από πρωτοβουλία της καγκελαρίου Μέρκελ, να ξεκινήσει μια διαφορετική διαδικασία και να δημιουργήσει μια διεθνή πλατφόρμα και να επιβάλλει την πρωτοκαθεδρία του ΟΗΕ και τη διαδικασία του ΟΗΕ. Μια διαδικασία που η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα στήριζε, πάντα στήριζε τον ΟΗΕ. Αυτό τι πλεονέκτημα έχει. Ότι όλες οι υπόλοιπε πρωτοβουλίε εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο του Βερολίνου. Γι' αυτό ο ύπατο εκπρόσωπος είπε από την αρχή ότι παρακολουθεί το θέμα της Λιβύης από την αρχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με τη Λιβύη από την αρχή και θέλει να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θέλουμε να εστιάσουμε στα δύο βασικά κατεπήγοντα. Το Βερολίνο, ε, από το Βερολίνο προέκυψε με μακρά δήλωση, με 54 σημεία αν την απατώμε, με, πολύ, με πολλά θέματα. Από τα πιο επίγοντα, ε, εφαρμογή του εμπάργου των όπλων και κατάπαυση του πυρός. Αυτά είναι τα πιο επίγοντα. Εκεί εστιάσαμε την προσοχή μας, αυτά τα δύο σημεία. Ο ύπατος εκπρόσωπος ζήτησε επίσης στις 10 Ιανουαρίου να γίνει μια έκτακτη συνάντηση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και μάλιστα μίλησε και για συγκεκριμένες επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στηρίξει την, τον ΟΗΕ και τη διαδικασία του Βερολίνου. Δεν ήταν εύκολα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλές ευαισθησίες, αλλά χθε ελήφθη ομόφωνα αυτή η απόφαση για να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση στη Μεσόγειο. με δορυφόρους με εναέρια κάλυψη και με θαλάσσια συνιστόσα. Κάτι διαφορετικό σε σχέση με τη Σοφία. Η Σοφία υποτίθεται θα τέλειωνε μέσα Μαρτίου. Και θα τελειώσει μέσα Μαρτίου. Τώρα με αυτή την επιχειρήση θα έχουμε μια νέα εντολή. Και θα έχουμε μια εστίαση για την, στην εφαρμογή του εμπάργου όπλων των ΟΗΕ. Η ιδέα ποια είναι. Να ληφθεί μια απόφαση μέχρι το επόμενο Συμβούλιο, δηλαδή μέχρι τις 23 Μαρτίου. Τώρα, τα στοιχεία της αποστολής θα θεσπιστούν, προφανώς, στην πορεία και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις διάφορες ευαισθησίες, αλλά υπάρχει πολιτική βούληση και το ομόφωνο μήνυμα των 27 κρατών μελών. Εν συνεχεία, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γενικά σε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της διαδικασίας του Βερολίνου. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Είμαστε δραστήριοι σε διάφορους τομείς με την ε, στήριξη του ΟΗΕ, οικονομική στήριξη, παραδείγματο χάρη που θα θέλαμε να δώσουμε στον ΟΗΕ στη Γενέβη, μα ενθαρρύνει πάρα πολύ Κάτι που μας φαινόταν αδύνατον στην αρχή. Χαιρόμαστε που καταφέραμε δηλαδή τώρα να φέρουμε τις δύο μεριές σε ένα κοινό τραπέζι και να συνεχίσουμε τη διαδικασία 5 συν 5 για το πώς θα εφαρμοστεί η κατάπαυση του πυρός. Θέλω να χαιρετήσω εδώ την προσπάθεια της Στέφανη και τις προσπάθειες του στρατηγού Σαλαμέ. Συγγνώμη, του ειδικού εκπροσώπου του ΟΗΕ Σαλαμέ. Η Στέφανη μας είπε ποια είναι η κατάσταση επιτόπου, η οποία δεν είναι ενθαρρυντική Άκουσα κάποιους να λένε ότι από τη μία έχουμε τον άξονα του Βερολίνου και από την άλλη έχουμε την πραγματικότητα επιτόπου. Παραμένουμε όμως πεπισμένοι ότι το Βερολίνο δημιούργησε μία ορμή. Θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί για να δούμε τα αποτελέσματα της διαδικασίας του Βερολίνου. Όπως και ο ΙΕ, και εμείς είμαστε ικανοποιημένοι που το Συμβούλιο Γενική Ασφαλείας κατάφερε την περασμένη εβδομάδα να υιοθετήσει το ψήφισμα, ένα ψήφισμα, το οποίο ζητάει την κατάπαυση του πυρός και που καταδικάζει τις πολλές και πολύπλευρες παραβιάσεις του εμπαργόπλων. Αυτό που συμβαίνει στη Γενέβη είναι θαρρυντικό και θέλουμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Το πρώτο μήνυμα που δώσαμε το έδωσε στη διάσκεψη του μονάχου ο ύπατος εκπρόσωπος Μπορέλ. Εδώ στις Βρυξέλλες θα διοργανώσουμε την τρίτη συνάντηση δημοσίων υπαλλήλων για το μηχανισμό follow-up. Η πρώτη συνάντηση έγινε την Κυριακή στο Μόναχο αυτού του επίπεδου, όπου έγινε μία συζήτηση και μία απογραφή των διαφόρων προβλημάτων. Τώρα, ε, ώρα ερωτήσεων, κύριο Γκάλα έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και για τις πληροφορίες ε, από τη Γενέβη και από εδώ στις Βρυξέλλες. Ε, έχω εκνευριστεί τώρα λίγο που εδώ στην ημερήσια διάταξη λέγεται μετά από την διάσκεψη στο Βερολίνο και εφαρμογή του εμπάργου στη Λιβύη. Έχουμε ακούσει για την κατάσταση του εμπάργου πολλά δεν ξέρω, εδώ οι εκπρόσωποι μπορούν να μας δώσουν κάποια εκτίμηση όσον αφορά την εφαρμογή του όπλων. Διότι εγώ έχω, ακούω πολλά ερωτηματικά. Ε, ναι, μεν αποφασίστηκε, αλλά οι ερωτήσεις μου είναι πολύ συγκεκριμένες. Στην περιοχή που βλέπουμε πάντα στους χάρτες, ε, αν με τι άλλο, είναι αποκλειστικές περιοχές που θέλουμε να ελέγχουμε. Τι γίνεται με τα πλοία που έρχονται από τη Ρωσία και από την Τουρκία, ελέγχονται και αυτά. Αυτοί είναι οι δύο βασικότεροι ε, που παραδίδουν όπλα. Τι γίνεται με τα άλλα ενδεχομένως ιδιωτικά πλοία ε, αυτοί οι Ρώσοι στρατιώτες, ε, οι ρωσικές παραδόσεις, τι έχει συμφωνηθεί με την Αίγυπτο για τα όπλα που έρχονται ε, με χερσαία μέσα από την Αίγυπτο. Υπάρχει έλεγχος των αεροδρομίων στη Βεγγάζη, στην Τρίπολη ή των πολλοστρατιωτικών αεροδρομίων. Όλα αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη. Τι γίνεται με τα κράτη του κόλπου που επίσης έχουν παραδώσει όπλα. Ποια είναι η δέσμευση αυτή τη στιγμή που επικυρώθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας ε, για όλους αυτούς που παραδίδουν όπλα. Και με ποια συγκεκριμένα ε, ε, πλοία ή με ποια μέσα θα βρεθούμε εμείς να ελέγχουμε τα πράγματα επί Τι συμφωνήθηκε ουσιαστικά. ούτως ώστε να υλοποιηθεί μια εκεχηρία, να πάψουν να μπαίνουν άλλα όπλα. υπάρχουν πολλά ακόμα ερωτηματικά όσον αφορά ε, το εμπαργκό παρά ε, πιστευτές απαντήσεις. Ε, μπορείτε να μας τα απαντήσετε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πέτερς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους διαμιλητές για τις πληροφορίες τους. Τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, η εμπλοκή της Τουρκίας στη Λιβύη με την αποστολή στρατευμάτων. Τι επίπτωση έχει αυτή η απόφαση της Τουρκίας. Πώς επηρέασε την ε, διάσκεψη του Βερολίνου. Δεύτερη ερώτηση. Το εμπάργκο όπλων. Εύκολο είναι το δηλώσεις. Το, αλλά πιο δύσκολο είναι να ελέγξεις το κατά πόσον υπάρχει και εφαρμόζεται το εμπάργκο όπλων. Υπάρχουν ήδη πολλά όπλα στη Λιβύη. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξή. Ο έλεγχο. Πώ εξασφαλίζεται. Τρίτον, μπορεί να υπάρξει τραπεζική κρίση στη Λιβύη. Το άκουσα και το κατάλαβα. Ποια είναι τα πρακτικά βήματα που μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε την τραπεζική κρίση. Και αυτή τη στιγμή σε ενσκύψει η, εγκύψει συγγνώμη, τραπεζική κρίση, τι κάνουμε τότε. Κύριε Νόρμαν, ευχαριστώ και τους δύο μιλητές για την πλήρη περιγραφή της κατάστασης στη Λιβύη. Συμφωνώ με τις ανησυχίες του κύριου Γκάλερ, ότι προσπαθούμε να καταλάβουμε λιγάκι ε, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε την, το εμπάργκο όπλων. Θέλω να σε ρωτήσω συγκεκριμένα, σε ποιο βαθμό καταλαβαίνετε τους δρόμους που χρησιμοποιούν οι δηλαδή λαθρέμποροι όπλων για να φέρουν όπλα μέσα στην χώρα. Λαμβάνουμε υπόψη μας το ποιοι είναι αυτοί οι δρόμοι. Παραδείγματος χάρη, τα περισσότερα όπλα έρχονται από την, από, για τις χερσαίες, οδού. Άρα τι γίνεται με τα χερσαία σύνορα. Δεύτερον, αυτή η νέα αποστολή θα παρακολουθεί ποιο παραβιάζει το εμπάρκο όπλων ή θα εμποδίσουμε τον κόσμο να φέρνει όπλα μέσα στη Λιβύη, γιατί δεν είναι καθόλου το ίδιο αυτό το πράγμα. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Γιατί δεν κατάλαβα τελικά ποιο είναι ο στόχο τη αποστολή. Τρίτον, πέρα από την παρακολούθηση και ίσω και, και την παρεμπόδιση, θα ονοματίζουμε και θα στυλιτεύουμε αυτούς που παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων και θα τους επιβάλλουμε κυρώσεις. Θα συγκεντρώνουμε πληροφορίες για τα ευρωπαϊκά όπλα, ευρωπαϊκά παραγόμενα όπλα, ας πούμε, που τελικά με κάποιον τρόπο βρίσκουν το δρόμο και μπαίνουν στη Λιβύη, μέσω του Κατάρ κτλ. Και τελευταία ερώτηση. Για τη δουλειά που θα κάνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Πότε θα αρχίσει να είναι επιχειρησιακή η αποστολή, τι χρονοδιάγραμμα έχουμε. Uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την κυρία Williams και την κυρία Τζίλη για την παρουσία τους εδώ σήμερα. Είναι ζωφερή κατάσταση βεβαίω στη Λιβύη και νομίζω ότι ήταν και σοφή η απόφαση που ελήφθη χθε. Είναι και ένα απαραίτητο βήμα αν ε, παίρνουμε και του εαυτού μα σοβαρά και πραγματικά θέλουμε να έχουμε κάποια επιρροή στη Λιβύη. Χρειαζόμαστε αυτό το πρώτο βήμα και ίσως και η ερώτηση προς την κυρία Βίλιαμ, γιατί είπατε ότι αυτό είναι ένα καλό και ένα πρώτο απαραίτητο βήμα αλλά ποια είναι η απόψη σα για το δεύτερο βήμα, τι πρέπει να κάνουμε. Και την ίδια ερώτηση αν ε, μπορούμε να έχουμε για παράδειγμα ένα ε, όργανο Παρακολούθηση Υπάρχει μια ναυτική αποστολή, αλλά τι γίνεται με τα χερσαία σύνορα. Υπάρχει, ναι, υπάρχει μια μεγάλη έκταση χερσαίων σύνορων ε, στη Λιβύη. Και τι κάνουμε για να παρακολουθήσουμε εκεί την κατάσταση. Τελειώσαμε τι ερωτήσει. Θα κάνω κι εγώ μια τελευταία ε, ερώτηση. Λίγο πριν τη σύνοδο του Βερολίνου, υπογράφηκε ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης της Λιβύης και της Τουρκίας, το οποίο έχει στρατιωτική, ένα πλαίσιο στρατιωτικής συνεργασίας ε, Τρίπολης-Άγκυρας, αλλά έχει ένα άλλο πλαίσιο, το οποίο είναι η συμφωνία ε, για τις ΑΟΣ των δύο χωρών, οι οποίε αυτή η συμφωνία παραβιάζει πλήρως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Εσείς από τη δικιά σας πλευρά πώς βλέπετε αυτή τη συμφωνία να εξελίσσεται μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης αυτά τα δύο θέματα, το ένα αφορά την Ελλάδα, το άλλο αφορά την ε, τον εμφύλιο της Λιβύης το επόμενο διάστημα. Four minutes each. If you got a time. Miss Williams, please. For four minutes. Uh, sure. Ναι, ναι. Νομίζω ότι θα αναφέρω τα θέματα που αφορούν την ε, εντολή των τι κάνει τα Έθνη. Όσον αφορά τις παραβιάσεις του εμπάργου όπλων ε, και το εμπάργο όπλων, όπως σας είπα, εγώ πιστεύω ότι η απόφαση που ελήφθη εχθές ε, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ήταν ένα θετικό πρώτο βήμα διότι δεν έχουν ε, υπάρξει πολλά θέματα παρακολούθησης ε, του εμπάργου όπλων καθόλου και ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες ε, παραβιάσεις. Θα ήθελα να σας παραπέμψω στις εξαντλητικές εκθέσεις των πάνελ εμπειρογνωμόνων τα τελευταία χρόνια, τα, οι οποίες αναφέρουν διεξοδικά και τις χώρες οι οποίες έχουν παραβιάσει το εμπάργο όπλων. Δεν υπάρχει κάποια πραγματική παρακολούθηση δεν έχουν επιβληθεί κυρώσει στις χώρες αυτές και δεν υπάρχει καμία λογοδοσία. Πρέπει λοιπόν να σταματήσει αυτή η ψευδέστηση των ξένων μαχητών, να σταματήσει να υπάρχει αυτή η ζωή ε, ε, όπλων ε, και θα το χρειαστούμε αυτό αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε ε, μια συνολική και διαρκείας κατάπαυση πυρός. Και φυσικά υπάρχουν θέματα και από τους γείτονες της Λιβύης, οι οποίοι πλήττονται ε, από την κρίση στην περιοχή και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγματι, πολλά πράγματα περνούν στη Λιβύη από ξηράς, ε, αλλά και από τη θάλασσα και από αέρος, επομένως πρέπει να υπάρχει κάποιο συνολικός μηχανισμός παρακολούθησης. Όσον αφορά τις χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή παρεμβαίνουν στη Λιβύη, το μήνυμα θα πρέπει να είναι ε, κάτω τα χέρια από τη Λιβύη, τις αρνητικές επεμβάσεις σας θα πρέπει να τις μετατρέψετε σε θετικές παρεμβάσεις και θα πρέπει να ε, έχουμε μια συνολική και μόνιμη λύση στο πρόβλημα της Λιβύης. Είναι μια χώρα η οποία βιώνει χάος και κρίση εδώ και μια χρόνια. Και εμείς πιστεύουμε και είμαστε πολύ ευγνώμονες για τα όσα επιτεύχθηκαν ε, στο Βερολίνο, ότι τα συμπεράσματα του Βερολίνου και το επιχειρησιακό σχέδιο Άσμαλ και το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών μπορούν να έχουν τα ουσιαστικά στοιχεία του προβλήματος της Λιβύης και κινούμαστε παράλληλα σε αυτές τις τρεις οδούς, το καθένα δημιουργεί εμπιστοσύνη για, τον, για την άλλη οδό. Και επομένω, θεωρούμε ότι αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ε, όσα υπέρφου, υφέρπουν σε αυτή τη ε, σύγκρουση διαρκείας. Ευχαριστώ πολύ. Yes, thank you. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα υπόλοιπα. Όσον αφορά τις σαφείς προϋποθέσεις. Ειλικρινά δεν έχω κάποια απάντηση. Ε, αποφάσεις ε, λαμβλήθηκαν χθες ε, βάσει μιας πολιτικής συμφωνίας μεταξύ των 27. Τώρα θα ξεκινήσουν άμεσα οι συνομιλίες για να καθοριστούν οι προποθέσεις. Δεν ξέρω ποια ακριβώς θα είναι η εντολή για την αποστολή. Θα αναφέρει πιθανότητα τους γενικούς στόχους. Θα αφορά παρακολούθηση, επιβολή. Θέλουμε να είμαστε λίγο ρεαλιστές, ρεαλιστικοί. Θα είναι περισσότερο παρακολούθηση παρά επιβολή. Αλλά πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν και οι επαφές με τα Ηνωμένα Έθνη σε αυτό το επίπεδο. Και το πώς θα υπάρξει μια άμεση επαφή με το πάνελ εμπειρογνωμόνων το οποίο αναφέρθηκε. Αυτοί πολύ περισσότερο από εμάς ε, έχουν επιφορτιστεί με το καθήκον του να κατονομάζουν τους ε, υπευθύνους και το κάνουν ε, με πολύ σαφή τρόπο γιατί είναι πολλαπλές οι παραβιάσεις από πολλές πλευρές τα ονόματα που έχουμε ακούσει είναι σωστά. Υπάρχει το ενδεχόμενο κυρώσεων μόνο που όταν μιλάμε για διασκέψεις τα πράγματα περιπλέκονται. Είναι πιο περιπλοκό σε ένα τέτοιο πλαίσιο να επιβάλλουμε κυρώσεις. Επίσης όμως έχουμε επενδύσει σε μια ευρεία διπλωματική προσπάθεια για να επικοινωνήσουμε με τις χώρες που ξέρουμε ότι θα αποτελέσει το κλειδί για να επιληθεί η κρίση στη Λιβύη. Ναι, πράγματι παρακολουθούμε τη θάλασσα, επειδή ρωτήσατε, αλλά όπλα φτάνουν ε, κατά κύριο λόγο με χερσαία μέσα και ένα το να έχουμε πλοία στη θάλασσα σημαίνει και τη χρήση ραντάρ. Οπότε, πολύ συγκεκριμένα δημοσιονομικά, είναι διανόητο να μπορούμε να εφαρμόσουμε μια τέτοια, να κρατήσουμε μια τέτοια ε, αποστολή. Χερσαία, για παράδειγμα, στα σύνορα μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης. Είναι τεράστια χώρα η Λιβύη. Είναι αδύνατο για μας κάτι τέτοιο. Αλλά οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες έχουν ε, πιστεί για την αποτρεπτική δυνατότητα που προσφέρει η χρήση θαλάσσιων μεσών σε συνδυασμό με δορυφορικά μέσα και για τη λαθρεμπορία και για την εμπορία ανθρώπων. Για το μνημονίο συνεννόησης μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας δεν έχω να πω κάτι που δεν έχει υποθεί ακόμα στο ανώτατο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 12 Δεκεμβρίου στο Ευρω... Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μήνυμα ήταν σαφές στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ειδικότερα στο ε, μνημόνιο συνεννόησης για τους περιορισμούς, για τα κυριαρχά δικαιώματα των κρατών μελών, ε, για τη μη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας ε, και για την μη δυνατότητα νομικών αποτελεσμάτων. Ευχαριστούμε.